Κυρία Ματέρα, δεν είμαι ικανοποιημένη. Ούτε εγώ. Ανέμενα περισσότερη, μεγαλύτερη πρόοδο όταν ανέλαβα ως αρμόδια επίτροπος για την ισότητα των φύλων. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο κινούμεθα. Κάποιος χαρακτήρισε τους καιρούς που ζούμε καιρούς αγωνίας. Βλέπουμε πολλές ανασφάλειες, εκνευρισμό στην κοινωνία μας, αγωνία και όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα ο κόσμος τίνει περισσότερο να αναδιπλώνεται ε, σε παλιές σε παραδοσιακές δομές και νοοτροπίες που έχουν αποδείξει την αξία τους στο παρελθόν. Αυτή η καιρή λοιπόν η δύσκολη δεν είναι ευνοϊκή για νέες τάσεις και ε, για νέες έννοιες και αντιλήψεις που θα γίνουν αποδεκτές από την ευρύτερη κοινωνία. Γι' αυτό ε, λέμε ότι είναι μικρή πρόοδος και τα αποτελέσματα, αλλά θέλω να το αιτιολογήσω. Γι' αυτό είναι τόσο μικρή η πρόοδος. Πρόσφατα κάποια κυβέρνηση δεν είχε καθόλου γυναίκε στη σύνθεση της Κυβέρνηση Ουγγαρία. Τώρα είπε η κυρία Μπλανκεβιτσούτε ότι στην ε, λιθουανική κυβέρνηση δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Και στις χώρες αυτές οι γυναίκες φαίνεται να διαφορούν. Είναι πολύ χλιαρές οι αντιδράσεις. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες, τα κράτη-μέλη να εκφράζονται και να διαμαρτύρονται, να λένε ε, ε, ότι δεν τους αρέσει αυτή η αδικία να μην συμμετέχει καμία γυναίκα στην κυβέρνηση. Ας εμπιστευτούμε ε, τους πολίτες. Θα εκφράσουν εκείνοι τις απόψεις τους, θα πούν πώς θέλουν να ζουν. Εγώ ανέκαθεν ήμουν κατά της νομοθετικής επιβολής της των ρόλων ναι, της, το πώς ε, θα ε, συνδυάζει κανείς τον επαγγελματικό με τον ιδιωτικό βίο, άνδρες και γυναίκες. Αυτό δεν επιβάλλεται δια νόμου. Ε, εκεί θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, σε αυτό το δρόμο, να δίνει ευκαιρίες, να ενισχύει την ισότητα, να μην ανέχεται τις διακρίσεις. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν και θα πρέπει να τα τονίσουμε, αλλά χωρίς να επιβάλλει δια νόμου. Με έξυπνη πολιτική όπου χρειάζεται να έχουμε νομοθεσία, αλλά ε, και μάλιστα η κείμενη νομοθεσία εδώ ε, λειτουργεί πολύ καλά. Ε, με συνειδητοποίηση, χρηματοδότηση, εκπαίδευση κτλ. Το δεύτερο σχόλιο, κύριε Γιούρεκ, Ξέρω τι είπαμε για τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Σεβόμαστε το δικαίωμα των κυρίαρχων κρατών να την κυρώσουν ή να μην την κυρώσουν. Θέλω μόνο να επαναλάβω ότι θα συνεχίσω να εξηγώ ε, για να διαλύονται κάποιες παρεξηγήσεις και παραπλανητικά επιχειρήματα που κυκλοφορούν σχετικά με την ερμηνεία της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται και τι είναι και τι δεν είναι η Σύμβαση. Είδατε κύριε Πρόεδρε, ήθελα να μιλήσω λίγο, αλλά δεν τα κατάφερα. Πολύ ωραία τα καταφέρατε, λέει ο πρόεδρο. Ε, δεν ακρηγορήσατε. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας και για την παρουσία σας. Ε, κλείνει εδώ η συζήτηση. Έχω λάβει δύο προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί αυτή. Μία από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και μία ε, πρόταση από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολιτικέ προκλήσει και στατηγικέ για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συνοσυρωτήτων. Εκ των συντακτών, το λόγο τώρα έχει η κυρία Αγιούτο. Παρακαλώ, για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Κάθε μέρα χιλιάδες γυναίκες αντιμετωπίζουν τη δική τους τη μάχη κατά της μάστιγας του αιώνα, του καρκίνου και το κάνουν αυτό ενώ με κουράγιο προσπαθούν να φροντίσουν παράλληλα και τις οικογένειές τους, ενώ προσπαθούν παράλληλα να διατηρήσουν και την εργασία τους. Για τις γυναίκες λοιπόν αυτές, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, θέλουμε μια πιο εύκολη και προσιτή πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις και στη θεραπεία. Τα στατιστικά δεδομένα της Eurostat μας ανησυχούν πάρα πολύ. Ένα στους τρεις Ευρωπαίους αναπτύσσει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του και περίπου 600.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους και 90.000 συγκεκριμένα από τον καρκίνο του μαστού, ενώ υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που παρουσιάζουν καρκίνο τη μήτρα ή καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα. Ο καρκίνο πλήττει του πάντε, γυναίκε, άντρε, αλλά ακόμα και τα παιδιά. Αλλά ξέρετε ότι όταν ο καρκίνο πλήττει τι γυναίκε, πλήττει ουσιαστικά τα γυναικεία χαρακτηριστικά των γυναικών. Δεν μα μας αφαιρεί ουσιαστικά τα τμήματα αυτά του σώματο, μα κάνουν να αισθανόμαστε γυναίκε, όπω το παραγωγικό σύστημα ή ο Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ψυχολογικές επιπτώσεις μετά την εμφάνιση του καρκίνου, ακόμα και μετά τη θεραπεία του καρκίνου. Σε σχέση με τα στατιστικά αυτά δεδομένα που έχουμε για τους πάρα πολλούς θανάτους, έχουμε ευτυχώς και πολλές γυναίκες οι οποίες καταφέρνουν να επιβιώσουν. Πάνω από το 80% των Ευρωπαίων γυναικών που έχει πληγεί από τον καρκίνο του μαστού καταφέρνουν τελικά να επιβιώσουν. Και είναι ακριβώς αυτές τις γυναίκες που πρέπει να προστατεύσουμε. Αυτές και τις οικογένειές τους. Μετά την ασθένεια συγκεκριμένα, η ζωή τους αλλάζει με τρόπο ριζικό είτε εξαιτία των πολύ έντονων ε, θεραπείων που πρέπει να κάνουν, όπω χημιθεραπεία ή ακτινοβολίε που πρέπει να δεχθούν, ή ακριβώ επειδή πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε χειρουργικέ επεμβάσει που έχουν επιπτώσει όχι μόνο σωματικέ. Α μην ξεχνάμε πώ αισθάνεται μια γυναίκα μετά από μια ιστεροκτομή ή μια μαστεκτομή. Οι επιπτώσει είναι όχι μόνο σωματικέ αλλά και ψυχολογικέ. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού με τα κράτη-μέλη να υπάρχουν συγκεκριμένε πολιτικέ που να λαμβάνουν υπόψη όλε αυτέ τι διαφορετικέ πτυχέ τη έκφανση του καρκίνου, όλων αυτών των σημαντικών επιπτώσεων που κρύβονται πίσω από τον καρκίνο. Τρία σημαντικά ζητήματα θα ήθελα καταρχάς να τονίσω. Πρώτον, πρόληψη και παρακολούθηση και πρόσβαση στι διαγνωστικές εργασίες. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου έχει να κάνει πολύ συχνά με το ότι ε, ο καρκίνος εντοπίζεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Επομένω, οποιαδήποτε θεραπεία στο στάδιο αυτό είναι πολλές φορές μάταιη. Καταλαβαίνετε ότι αν η διάγνωση γίνει πολύ πιο νωρίς, το ποσοστό επιβίωσης είναι πάρα πολύ πιο υψηλό. Θα πρέπει λοιπόν και από οικονομικής πλευράς να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών στις απαραίτητες εξετάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος προσυμπτωματικός έλεγχος, ο οποίος να είναι διαθέσιμες για όλες τις γυναίκες. Ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές γυναίκες χρειάζονται να καταβάλουν πολύ σημαντικά ποσά ή περιμένουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, ε, διαγνωστικές εξετάσεις. Δεύτερον, οι συγκεκριμένες θεραπείες που θα πρέπει να γίνουν των ασθενούν οι γυναίκες. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε καρκίνους που έχουν να κάνουν με γυναικεία όργανα όπω ο μαστός ή η μήτρα. Καταλαβαίνετε ότι οι θεραπείε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονό ότι έχουμε να κάνουμε με τμήματα του σώματο που έχουν, να που έχουν άμεση σχέση κάνουν ουσιαστικά τι γυναίκε να αισθάνονται γυναίκε. Νομίζω λοιπόν ότι πέρα από την λειτουργική αισθητική πλευρά υπάρχει και μια πολύ έντονη ψυχολογική πτυχή. Και τρίτο σημαντικό ζήτημα, η ψυχολογική πλευρά και το ζήτημα της υποστήριξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε καταλήλως τις γυναίκες που μαστίζονται από τον καρκίνο. Αυτή τη στιγμή μια γυναίκα ξεκινάει μια μάχη κατά τον καρκίνο και χρειάζεται ουσιαστικά να κάνει επεμβάσει και χρειάζεται ουσιαστικά να στερηθεί τα τμήματα εκείνου του σώματό τη που συνδέονται άμεσα με τη γυναικεία τη φύση και πολλέ φορέ οι επεμβάσει αυτέ είναι μη αναστρέψιμε. Καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση αυτή οι ψυχολογικέ επιπτώσει ακόμα και κατά το μεταχειρητικό στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπετε μια ψυχολογική υποστήριξη για όλε αυτέ τι γυναίκε. Το να αφήσουμε μόνε του τι γυναίκε αυτέ ουσιαστικά ισοδυναμεί με το θα ε, θα καταστήσουμε τη ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Θα πρέπει οι γυναίκες αυτές εντελώς ε, μόνες να χρειαστεί να τα βγάλουν πέρα, φέροντας ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Ένα κοινό πρόγραμμα προσυμπτωματικών ελέγχων που ουσιαστικά να ε, διέπεται από μια συγκεκριμένη υποδομή υγειονομική περίθαλψη. Σας ευχαριστούμε. Ο Επίτροπο τώρα έχει το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εξώτημα μέλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Επομένω, επιτρέψτε μου ε, και δώστε μου λίγο περισσότερο χρόνο για να απαντήσω ολόπλευρα σε αυτό το πολύ λεπτό και ιδιαίτερο ζήτημα. Ευχαριστώ ε, την κυρία Γιούτο, την αγαπητή Ντανιέλα, που έθιξε αυτό το ζήτημα ε, για τις ασθένειες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τα στατιστικά καταμαρτυρούν μια τρομερή κατάσταση. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου. Πάνω από 580.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πέρσι. Σχεδόν 4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις αναμένονται μόνο για φέτος. Όμως αυτό το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα στατιστικά στοιχεία. Ο καρκίνος επλήττει τις ε, οικογένειες, ε, τις οικονομίες ε, και ούτω καθεξής. Από το πρώτο πρόγραμμα κατά του καρκίνου το 1980 η επιστήμη, η έρευνα και η δημόσια πολιτική έχουν οδηγήσει σε νέες πρωτοβουλίες, καλύτερη ε, διάγνωση, καλύτερη πρόληψη και καλύτερη θεραπεία του καρκίνου. Έχουμε πετύχει πολλά λοιπόν από κοινού. Η νομοθεσία για τον καπνό ε, και για άλλους ε, τομείς η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και των εθνικών προγραμμάτων ε, κατά του καρκίνου είναι απτά παραδείγματα ευρωπαϊκών επιτευμάτων. Τώρα, για τα ερωτήματά σας. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, να τονίσω ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ήδη συνεργάζονται σε ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια κατά του καρκίνου προκειμένου οι ασθενείς ε, ε, να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα υψηλής ποιότητας. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τους βασικούς ε, παράγοντες, τους καρκινογόνους παράγοντες, να έχουμε σωστή πρόληψη και πρόημη διάγνωση για να καταπολεμήσουμε ειδικούς, ειδικές μορφές καρκίνου. Αυτό έχει να κάνει και με τις Ευρωπαϊκές Κατηγορίες Γραμμές του 2017. που περιλαμβάνουν και μια σύσταση για τους διαγνωστικούς ελέγχους, την άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ποιοτική θεραπεία και ε, στήριξη και μετά τη θεραπεία ε, και σε ό,τι αφορά τους ε, όσους ξεπερνούν και κατανικούν τον καρκίνο, τη σωστή υποστήριξή του. Βλέπουμε ότι Έχουμε και νέου δείκτε που εκφράζουν με ποσοτικό τρόπο ε, τα στοιχεία ανά την Ευρώπη. Αυτό επιτρέπει την χρήση ε, συγκεκριμένων προτύπων ε, θνησιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τι προσπάθειε των μελών και στον εμβολιασμό και σε ό,τι αφορά το, την υπατήτηδα και τον HPV που προκαλεί καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στις γυναίκες. Και σας ζητώ ε, να μας βοηθήσετε να καταπολεμήσουμε ε, τη διστακτικότητα που υπάρχει ε, απέναντι στα εμβόλια. Γιατί είναι σημαντικό ζήτημα. Γενικά υπάρχει σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα περιστατικά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Σχεδόν, όλες, σχεδόν όλα τα κρατημέλη έχουν σχέδια δράσης. Το καλύτερο θα ήταν να είναι όλα βέβαια αλλά πριν από 10 χρόνια ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έχει αυξηθεί ο ρυθμός των γυναικών ε, που ε, περνούν από διαγνωστικό έλεγχο και είναι δύσκολο βέβαια να δώσουμε κίνητρο ε, στους πολίτες να κάνουν αυτούς τους διαγνωστικούς ελέγχους. Αυτό έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στα ποσοστά επιβίωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Δεύτερον, αν η Επιτροπή προβλέπεται να ε, διαμορφώσει πρότυπα διαγνωστικού ελέγχου. Υπερθυμίσω ότι υπήρξε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο του μαστού. Και έτσι καταλήξαμε σε κατευθυντήριες γραμμές που καλύπτουν όλο τον κύκλο από τον διαγνωστικό έλεγχο μέχρι ε, την ε, ε, ε, τελική θεραπεία και ε, υποστήριξη στα τελικά στάδια του καρκίνου. Όμω, όλε αυτέ οι βέλτιστε πρακτικέ και οι συστάσει και οι πρωτοβουλίε θα πρέπει να μεταφραστούν σε απτέ ενέργειε και πρωτοβουλίε στα κρατη Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε τα κρατη για να υλοποιήσουν αυτέ τι προτάσει μα επιτόπου. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, προώθηση της υγείας ε, και για τις ε, μη μεταδοτικές ασθένειες. για να συμβουλεύσουμε τα κράτη-μέλη με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι μπορούν να κάνουν. Μπορούν να υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη που μπορούν να υλοποιηθούν και σε πιο μαζική κλίμακα. Και το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα Horizon Ευρώπη εισάγει την ε, έννοια των ε, Mission Driven Initiatives, συγκεκριμένων πρωτοβουλειών, λοιπόν, με βάση ευρύτερους στόχους. Τρίτο, κατά πόσο υπάρχει εκστρατεία ετοιμότητα. Εξαιρετική ερώτηση αυτή. Η πρόληψη είναι ακρογωνιαίο λήθο ε, τη προσπάθειά μα. Ξέρουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, αλλά πώ μπορούμε να την ε, επιτύχουμε στην Ευρώπη. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με κράτη-μέλη, τον ΠΟΗ και τη ε, Διεθνή η υπηρεσία οργάνωση έρευνα κατά του καρκίνου για να προωθήσουμε τον Ευρωπαϊκό ε, Κώδικα κατά του καρκίνου, που είναι πολύ απλό, κατανοητό ε, και ισχυρό. Για να περιορίσουμε, να ποιώσουμε με τον κίνδυνο ε, καρκίνου, έχουμε εστιάσει συγκεκριμένε πολιτικέ κατά του καπνού, υπέρ τη άσκηση, τη υγιεινή διατροφή. Πολύ απλά πράγματα, αλλά ισχυρά μηνύματα. Επιπλέον, ε, προωθούμε τα προγράμματα διαγνωστικού ελέγχου και του, κατά του καρκίνου, του τραχύλου της μήτρας και ε, προωθούμε όσο μπορούμε τον εμβολιασμό ε, για την υπατήτητα Β και τον HPV. Έτσι αυτό, είναι ένας, αυτό το πλαίσιο είναι ένας απλός και κατανοητός ε, τρόπος για να ε, διαδώσουμε αυτό το μήνυμα για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο του καρκίνου. Όμως πάλι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την διοργάνωση, για παράδειγμα, των ε, εκστρατιών ετοιμότητας για τον καρκίνο, αύξηση της ευαισθητοποίησης και της επίγνωσης ό,τι αφορά τα προγράμματα διαγνωστικού ελέγχου. Εγώ είδα μάλιστα σε ένα αεροπλάνο την αεροσυνοδό ε, που ενημέρωνε τις γυναίκες ότι να ορίστε μπορείτε να κάνετε τον προκαρκινικό διαγνωστικό έλεγχο. Υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα. Πρέπει να παραμείνει πολύ ψηλά ε, στην λίστα προτεραιοτήτων αυτό το θέμα και στον δημόσιο διάλογο. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε πετύχει και σημειώσει πρόοδο, όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Χρειαζόμαστε ε, την έρευνα και την καινοτομία για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των ε, ε, ασθενών. Πρέπει να συνεχίσουμε να προαγάγουμε υγιείς συνθήκες και επιλογές ζωής, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κανείς δεν εξετάζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τέλος, υπάρχει και ένα προεκλογικό μανιφέστο σχετικά με τον καρκίνο και το χαιρετίζω αυτό σαν πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την συνολική αυτή απάντηση και εξαντλητική. Παρακαλώ να τηρούμε το χρονογόρευσή μας, γιατί έχουμε ξοκύλει κάπως χρονικά. Κυρία Πετήρ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι τρομακτικό το γεγονός ότι το 1 τέταρτο όλων των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονται σε καρκίνο. Σύμφωνα με ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, η Κροατία, το πιο νέο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Ουγγαρία, είναι από τις 10 πρώτες χώρες σε ό,τι αφορά τους θανάτους από καρκίνο. Ε, αυτό είναι στοιχεία ε, από το αρμόδιο ε, ίδρυμα, ε, το 2018 σημειώθηκαν 2 εκατομμύρια νέοι, νέα κρούσματα περιστατικά καρκίνου του μαστού. Και μάλιστα πρώτο είναι το Βέλγιο, μετά το Λουξεμβούργο και μετά 100 χώρες από επιπολασμό. Οι ε, αρρώστιες δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν γνωρίζουν εθνικότητες κτλ. Είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα και όλες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνειδητοποίηση, μια εκστρατεία, να το καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες, να γίνονται ε, προσυμπτωματικοί έλεγχοι ε, σε όλες τις γυναίκες, χωρίς καμία εξαίρεση και στους άνδρες. Είναι κοινό ο αγώνας μας και χρειάζεται συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλό θα ήταν να έχουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια. Και να μην ξεχνάμε όμως ότι η αρμοδιότητα για την υγεία παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Ευχαριστώ για δύο μισή λεπτά η κυρία Μπόρζαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, κυρίως να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, τη συντάκτρια της ε, ερώτησης για το καταπληκτικό ψήφισμα, την κυρία Αγιούτο. Και ευχαριστώ που έφερε το θέμα αυτό. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο περίπου 1,3 ε, εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο, το 1 τέταρτο όλων των θανάτων. Από την άλλη, ο καρκίνος του μαστού ε, έχει ψηλό ποσοστό επιβίωσης, 80%. Βεβαίως, αν ανακαλυφθεί εγκαίρος. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα ελέγχων και προσυμπτωματικών για όλους και όλες. Χωρίς αποκλεισμούς από το σύστημα υγείας. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να έχει καθολική πρόσβαση και ίση πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες που χρειάζεται, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους διαγνωστικούς ελέγχους για την έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη και μετά ε, την χειρουργική επέμβαση, ανεξαρτήτως του που ζει. Ας πούμε, γυναίκες καρκινοπαθείς που ε, γίνονται καλά μπορεί να έχουν άλλες δυσκολίες ψυχολογικές και τα λοιπά όταν επιστρέφουν ε, στο σχολείο, στην οικογένεια, στη δουλειά τους. Είναι επίσης πολύ ε, προβληματικό να διατηρηθεί και η αναπαραγωγική υγεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Φυσικά μπορούμε να ζητάμε πάρα πολλά, αλλά αν δεν έχουμε τα απαραίτητα χρήματα δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Στις δικές μου τροπολογίες Έχω τονίσει ότι ε, πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στην έρευνα και μάλιστα στην έρευνα για όλα τα είδη καρκίνου. Θα πρέπει να αντιδράσουμε ε, σε αυτή την ανησυχητική διάκριση που ε, έχουμε και τη διαφορά στα νούμερα και στους θανάτους από καρκίνο στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Παρακαλώ να το κοιτάξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας πούμε, ε, ο καρκίνος των οθικών ή ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας οδηγεί σε περισσότερους θανάτους στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει και με ε, τη ζωή που κάνει ο καθένας και με την υποστήριξη από το ιατρικό σύστημα, το σύστημα υγείας και την οικογένεια. Έχουμε κάνει πολλές υποσχέσεις, αλλά δεν τις έχουμε υλοποιήσει. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Ζιτνάνσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς στη Σλοβακία έχουμε κάθε χρόνο 30.000 νέα περιστατικά καρκίνου. Είναι από τις πιο θανατηφόρες νόσους. Παρά το γεγονός αυτό, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που διαγνώσκονται με καρκίνο. Τα τελευταία χρόνια ε, δεν έχουμε ένα σωστό ε, ογκολογικό μητρό. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί και να αρχίσει από τώρα η σωστή συλλογή στοιχείων στατιστικών δεδομένων. Μετά από τόσες προσπάθειες γιατρών και ασθενών ε, έχει ε, αρχίσει ε, να γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντερού και του μαστού. Ε, στις ο καρκίνο του μαστού είναι ο πιο συχνό καρκίνο. Δυστυχώ, όμω διαγνώστηκε σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή τους άδικα 300 γυναίκε. Ε, ε, χαίρομαι λοιπόν για τις μαστογραφίες και τους άλλους ελέγχους. Ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εξετάσεις να γίνονται καλά στο κέντρα και θα πρέπει να σπάσει αυτός ο μύθος ότι βλάπτει δίθεν η μαστογραφία και είναι ε, ε, κακή. Είναι η μόνη μέθοδος για να ε, μπορέσει κανείς να διαγνώσει εγκαίρως τον καρκίνο του μαστού. Λίγα λεπτά χρειάζεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος στη ζωή μια γυναίκας, αλλά μπορεί να τη σώσει τη ζωή. Να μην φοβούνται οι γυναίκες και να κάνουν check-up και προληπτικούς ελέγχους. Ευχαριστώ για δυόμιση λεπτά η κυρία Βίρινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κάιτης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πολλές είναι οι προκλήσεις στις πολιτικές μας για να βελτιώνουμε τη ζωή των καρκινοπαθών γυναικών. Για μένα αυτά ξεκινούν από την πρόληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η ποιότητα του ε, διαγνωστικού ελέγχου που πρέπει να εναρμονιστεί σε όλη την Ευρώπη. Ε, όσο νωρίτερα γίνεται σε ομάδες κινδύνου ε, μπορεί να μειώσει ριζικά τον αριθμό των ασθενών. Η ποιότητα της ζωής τους επηρεάζεται πάρα πολύ από κάθε μορφή καρκίνου. Γι' αυτό οι γυναίκες θα πρέπει να καταπολεμούν τις αγωνίες, την ανορεξία, την αϊπνία, την κατάθλιψη και επίσης ε, μπορεί να έχουν και νωρίτερα εμεινόπαυση που σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορεί να μην γίνουν ποτέ μητέρες. Εξού και ε, η πρωτοβολία ε, κατά του καρκίνου του μαστού είναι κάτι που υποστηρίζω. Ε, πέρα από κομματικά σύνορα, πέρα από γεωγραφικά σύνορα των κρατών μελών μπορούμε να συνομιλήσουμε με ενεχομένους, με ενδιαφερομένους για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού επηρεάζει ανετικά και την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών ο καρκίνος. Γιατί μπορεί να απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε δε που χάνουν και τη δουλειά τους. Ακόμα και μετά την ίαση ε, υφίστανται τις συνέπειες οι ασθενείς. έξω και είμαι ε, στεναρή υποστηρίχθεια τη ε, πρωτοβουλία στο δικαίωμα στη λύθη Δηλαδή μετά την ίαση να μπορεί κανείς να κάνει ασφάλειες, ε, να παίρνει δάνεια, σαν να μην είχε ασθενήσει ποτέ. Χάρη στην έρευνα και την καινοτομία έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην πρόληψη του καρκίνου, στην αντιμετώπιση του και στη φροντίδα για τους καρκινοπαθείς. Άρα υποστηρίζω και εγώ το αίτημα για εναρμονισμένη ε, ευρωπαϊκή πολιτική κατά του καρκίνου στραμμένη προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε τούτη εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα τα εμπορικά συμφέροντα των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών και άλλων εταιριών που έχουν κάνει εμπόρευμα την υγεία να μπαίνουν εμπόδιο στην ε, παρακολούθηση από τις δημόσιες υπηρεσίες ε, τη υγεία των γυναικών και των ανδρών. Όπω λέει η διαμεσολαβήτρια και τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, είναι αδύνατο να κρύψουν ε, τις συνεδριάσεις με τα λόμπι ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και εδώ που σποσοράρουν διάφορες εκδηλώσεις οι εταιρείε αυτές. Ε, το είδαμε στα εμφυτεύματα μαστού από μια γαλλική εταιρεία που ήταν προβληματικά και το οποίο τα τελευταία χρόνια εμεί καταγγέλαμε συνέχεια. Και παρά αυτή την κατακραυγή και το σκάνδαλο ε, συνεχίζουν άλλοι κατασκευαστές χωρίς να προειδοποιούν ε, για ε, τη σιλικόνη και τι ανεπιθύμητες ε, ενέργειες έχει. Γι' αυτό και την άλλη εβδομάδα θα το ξαναδούμε στην Επιτροπή Αναφορών. Το ίδιο ισχύει και με τα αντικακενικά φάρμακα που χρειάζονται ισχυρό σύστημα υγείας, οπωσδήποτε καθολικό και δημόσιο και όσο γίνεται με περισσότερα χρήματα και πόρους και να σέβεται και την ιδιαιτερότητα του κάθε φύλου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην πρόληψη παρακολούθηση, θεραπεία και συνέχεια όπως είναι στο καρκίνο του μαστού. Στη συνέχεια τα κράτη-μέλη που εκτελούν και υλοποιούν τα μέτρα για τη δημόσια υγεία θα πρέπει να έχουν μια καθολική θεώρηση, όχι μόνο απαραίτητη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, αλλά και στον έλεγχο των ε, προϊόντων υψηλού κινδύνου θα πρέπει να αξιολογούν πώς αυτά επηρεάζουν την υγεία των γυναικών. Τέλος, και τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα χρήματα από τα διορθωτικά ταμεία και τα υπόλοιπα μέσα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επενδύουν στην έρευνα, την ανάπτυξη σε ειδικά ε, ιατρικά κέντρα και σε ειδικευμένο προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ. Um, θα ευχαριστούμε. Η κυρία Ριβαζή το η οποία απουσιάζει όμω, Επομένως περνάμε στον επόμενο μιλητή, την κυρία Κοσλόφσκα Ράτσεβιτς. Για ένα λεπτό, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Όλες αυτές οι ασθένειες που συνδέονται ουσιαστικά με τον πολιτισμό μας, με την σημερινή, με τον σημερινό τρόπο ζωής, έχουν να κάνουν σαφώς με συγκεκριμένε πτυχές της ζωής μας, όπως η ατμοσφαιρική ρήπανση, η ζωή της πόλης κτλ. Και οδηγούν ουσιαστικά σε πολλές διαφορετικές μορφές καρκίνου. Πέρα λοιπόν από την ιατρική βοήθεια χρειάζεται συγκεκριμένη δράση όσον αφορά την πολιτιστική στάση που διατηρούμε, όσον αφορά τον τρόπο που ζούμε τελικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε το ζήτημα αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που προτείνονται πολύ συγκεκριμένοι τρόποι για το πώ μπορούμε να αποτρέψουμε τον καρκίνο και πώ μπορούμε να τον θεραπεύσουμε αν τυχόν εμφανιστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, στο ψήφισμα αυτό ε, γίνεται μια έκκληση όντω σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική και προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω να ακολουθήσει την έκκληση αυτή. Χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική, χρειαζόμαστε κοινή χρηματοδότηση και χρειαζόμαστε πρόσβαση στα καλύτερα δυνατά πρότυπα αντιμετώπιση του καρκίνου, έτσι ώστε κάθε γυναίκα, είτε ζει στη Δυτική ή στην Ανατολική Ευρώπη, να έχει τι ίδιε ευκαιρίε να θεραπευτεί αν τυχόν εμφανίσει καρκίνο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Η κυρία Βυσνέσκα τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Ένα στους τρεις Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια της ζωής του θα αναπτύσσει καρκίνο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα από 1.300.000 χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο, 26 περίπου του πληθυσμού τα βασικά αίτια του καρκίνου, οι βασικές μορφές μάλλον του καρκίνου που αντιμετωπίσουν οι γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος της μήτρας, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες είναι ο πιο συχνός καρκίνος και οδηγεί πολύ συχνά στο θάνατο. Συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αποκλήσεις και διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ιδίω ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, όσον αφορά τα πρότυπα αντιμετώπιση του καρκίνου. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μειωθούν οι αποκλήσει αυτέ και να έχουμε μια κοινή πολιτική, να καταφέρουμε να προωθήσουμε πιο υγιείς μορφέ ζωή και θα πρέπει σαφώ να προωθήσουμε ω το δυνατόν περισσότερο τον πρεσοπτωματικό έλεγχο. Σα ευχαριστούμε κυρία Σόιντροβα. Έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν πραγματικά ότι ο καρκίνος σκοτών, 26% των θανάτων οφείλεται στον καρκίνο. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε ως κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο έχουν προωθηθεί και διάφορες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, ο οποίος αναφέρθηκε σε πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές και είπε ότι και ο ίδιος προσωπικά δεσμεύεται και προσιλώνεται στο στόχο αυτό καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο αυτό και ότι γνωρίζει ότι δρά υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών και υπέρ των γυναικών που πλήττονται από τον καρκίνο. Όσον αφορά τους καρκίνους των γυναικών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των καρκίνων αυτών είναι ο καρκίνο του μαστού. Η πρόληψη λοιπόν του καρκίνου του μαστού θα πρέπει να περιλαμβάνει την προώθηση ε, πιο υγιού τρόπου ζωή, πιο υγιεινή διατροφή και θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον απαραίτητο προσυμπτωματικό έλεγχο. Είναι σημαντικό να προωθηθούν ευρωπαϊκέ εκστρατείε που πραγματικά θα βοηθήσουν τη μείωση τη εμφάνιση του καρκίνου αυτού. Ο κύριο Τζάμι τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως ακούσαμε στην αρχή της συζήτησης, συζητάμε εδώ πέρα ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Στην Μάλτα έχουμε 2.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο, 900 θανάτους κάθε χρόνο έχουμε 350 καρκίνους στους 2.000 που είναι καρκίνοι του μαστού. Έχουμε καλά ποσοστά επιβίωσης, 78% πάνω δηλαδή από το κοινοτικό μεσόρο. Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διδραματίσει ο προσηματικός έλεγχος. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών και των πολιτών στον προσματικό έλεγχο αυτό. Δεν αρκεί να υπάρχει μόνο έλεγχο αυτό, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και από του Ευρωπαίου πολίτε. Ξέρετε ότι Είχαμε στο παρελθόν και την παρουσία διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων που ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μα μίλησαν για αυτέ τι μορφέ του καρκίνου. Θα πρέπει να προωθήσουμε επίση την έρευνα και την καινοτομία και θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωή και επίση και πιο ποιοτικά τρόφιμα. Σας ευχαριστούμε. 7 ομιλητές θέλουν να πάρουν το λόγο στα πλαίσια του Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο σε όλους τους ομιλητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Κυρία Ζαμπόρσκα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω και η κυρία Γιούτα και εγώ θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου ακόμα μένουν πολλά ακόμα να γίνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ε, να μεριμνήσουμε τόσο ώστε ε, ο πρώιμος προσυμπτωματικό έλεγχο και η σωστή αντιμετώπιση, η θεραπεία από κοινού και με την προώθηση γεϊνών επιλογών ζωής καθώ και τη πρόληψη, Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αποτελέσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο θα πρέπει να υλοποιείται και να γίνεται σεβαστό από όλα τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς ε, σήμερα αυτά δεν είναι ο κανόνας. Παραμένουν ε, διαφορές και ανισομέρειες μεταξύ ε, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης και σε ό,τι αφορά τον επιπολασμό και σε ό,τι αφορά τα ποσοστά θνησιμότητας για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά και για άλλες μορφές καρκίνου. Δεν γίνεται να αποδεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Ο καρκίνος δεν επιλέγει τα θύματα του με βάση το φύλλο τους. Γι' αυτό ε, υποστηρίζω και το ψήφισμα και τις ε, τροπολογίες της κυρίας Πετήρ. Η 4η Φεβρουαρίου ήταν η μέρα κατά του καρκίνου και ήταν μια δυνατότητα για εμάς να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για τι ευρωπαϊκέ οικογένειε. Ω ε, ευρωβουλευτή, έχω το καθήκον να εντοπίσω και να αναδείξω τομεί στους οποίου μπορεί ε, να έχει καλύτερα αποτελέσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την πρόληψη του καρκίνου και για τη στήριξη προ τα θύματα. Πρέπει λοιπόν να αναδείξω ε, τη δυστυχία των γυναικών που πλήττονται από καρκίνους που έχουν να κάνουν με βιομηχανικέ ουσίε και, στη, και στους κλάδους λοιπόν του καθαρισμού και τη ομορφιά, αν θέλετε, οι γυναίκε ε, εκτίθενται ε, σε καρκινογόνους παράγοντε. Οι πολιτικοί, λοιπόν, ανά την Ευρώπη πρέπει να εξετάσουν περισσότερο τι μπορούμε να κάνουμε για να προλαμβάνουμε αυτού του καρκίνου. Πρέπει οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενε να έχουν ε, πρόσβαση σε προστατευτικά μέτρα σε ό,τι αφορά τι ουσίε που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνες. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να αυξάνεται ο κίνδυνο καρκίνου για τι γυναίκε, μόνο και μόνο εξαιτία τη δουλειά που κάνουν. Ο Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο καρκίνος θερίζει και αυτό αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. 26% των θανάτων προέρχονται από τον καρκίνο. Για τις γυναίκες έχει αποδειχθεί και από τη συζήτηση αλλά και τις μελέτες ότι ο καρκίνος βασικά αφορά τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο της μήτρας και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και φυσικά είναι δυνατόν να υπάρξει πρόληψη και σε αυτό το στάδιο πρέπει να εστιάσουμε να έχουμε πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ για τις γυναίκες να υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας και μάλιστα χαμηλού κόστους διότι διαφορετικά υπάρχει απαγορευτική πρόσβαση προς την θεραπεία από την πλευρά των γυναικών και φυσικά στο επόμενο στάδιο είναι να υπάρξει ψυχολογική στήριξη διότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται ιδίως η θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να οδηγήσει το 78% των γυναικών σε επιβίωση αλλά χρειάζεται από εκεί και πέρα στήριξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο καρκίνος είναι μια αρρώστια που αφορά τόσο πολλές γυναίκες στην Ευρώπη που υποφέρουν και σωματικά και ψυχικά και ψυχολογικά. Ε, εμείς υποστηρίζουμε όλες αυτές τις γυναίκες και την οικογένειά τους. Ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθολικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας που δεν θα πρέπει να περικόπτονται λόγω λιτότητα. Στη χώρα μου 40.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ε, το, την Κυριακή για την ε, υγεία, τη δημόσια υγεία ε, και μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται μαστογραφία και να εντοπίζεται εγκαίρως το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο ε, κατά του ιού ε, που προκαλεί ε, καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. HPV. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Και τέτρα στις νέες γυναίκες και στα κορίτσια πρέπει να γίνεται πρόληψη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο, λέει ο κύριος Πόλτσακ. Ε, θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ πολύ αυτά που είπε ο Επίτροπος. Ε, όλοι ε, συζητούμε για τα αποθέματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη του καρκίνου. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη και ο τρόπος ζωής. Η Λουτσία Πέταβα από την Τσεχική Δημοκρατία διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στην ηλικία των 28 ετών και έγινε ηρωίδα πραγματικά στην Τσεχία γιατί δεν φοβήθηκε να το δηλώσει αυτό δημόσια και να το συζητήσει. Και είπε μην είστε ανόητες, πηγαίνετε και κάνετε ε, ελέγχους διαγνωστικούς και πραγματικά ενθάρρυνε χιλιάδες γυναίκες να προχωρήσουν σε check-up και σε τεστ PAP. Ε, δεν είναι λύση από μόνο το της αυτή αλλά θα πρέπει οι γυναίκες να πηγαίνουν να κάνουν αυτούς τους προδιαγνωστικούς ελέγχους. Είναι πραγματική η ιστορία αυτή από την ε, Τσεχική Δημοκρατία. Κυρία Καπεθόνου Ρουίθ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά ζουν χειρότερα ε, διαδηλώνουν ε, πολύ συχνά γιατί δεν καλύπτονται ιατρικά. Μία στις 8 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάθει καρκίνο. ενώ ε, από 30 μέχρι 90% είναι ο έλεγχος σε ηλικία 50 με 69 ετών οι μαστογραφίες κλπ. Υπάρχουν καρκίνοι που προκαλούν πολλές ζημιές, ε, ε, στηρότητα αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν η διάσταση του φύλου να μπει και στα προβλήματα και στα προγράμματα υγείας και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ηγηθεί σε αυτή τη συνολική προσέγγιση των ε, καρκίνων των γυναικών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έρευνα, τον προδιαγνωστικό ε, προσυμπτωματικό έλεγχο, ε, την θεραπεία και την αποθεραπεία. Ευχαριστώ η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Ακόμα και παρότι έχει περάσει η ώρα, Έχουμε τόσο πολλά κρούσματα καρκίνου και σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Η πολιτική μας ομάδα υποστηρίζει την Ένωση ε, κατά πολέμηση του καρκίνου και νομίζω ότι και ο κύριος Επίτροπος γνωρίζει τις ε, του. Ε, πρέπει σίγουρα να έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση. Δεν γίνεται να ανεχόμαστε πλέον αυτό το χάσμα μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί είναι ενιαίος ο αγώνας για την ισότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ε, στη θεραπεία. Ε, Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε σίγουρα την κατάσταση. Ευχαριστώ, ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα και παρακολούθησα τη συζήτηση αυτή και σας είμαι ευγνώμων για την ε, συνεισφορά σας. Σε ό,τι αφορά τις ε, ιατρικές συσκευές και τα εμφυτεύματα και τα λεφτά. Έχουμε σχετική ε, ε, οδηγία πλέον, να προχωρήσουμε. Είναι στα χέρια μας να ρυθμίσουμε αυτό το περιβάλλον, μια που μιλάμε για πολυεθνικές και τελικά εταιρείε. Κοιτάξτε, για τα καρκινογόνα έχουμε βάλει ε, στον κατάλογο και νέες ουσίες, πολλές. Όταν συζητούσαμε για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία καταπολέμηση του καπνίσματος, ε, ενδοκρινικοί διαταράκτες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ρυθμίσουμε πιο αυστηρά ε, τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Έχουμε κάνει πολλά μαζί τα τελευταία 4,5 χρόνια και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, για την πρόληψη του καρκίνου. Αυτή είναι η συλλογική απάντηση ε, στα διάφορα προγράμματα πλαίσιο έρευνας η Ένωση έχει χρηματοδοτήσει τα προγράμματα αυτά από το 2007 για την πρόληψη με 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, κάντε τους υπολογισμούς, προχωρούμε. 440 εκατομμύρια έχουμε ψηφίσει τα τελευταία 10 χρόνια για τον καρκίνο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τον καρκίνο του μαστού ε, και τον καρκίνο του γεννητικού συστήματος. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε σύσταση για να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο σύστημα που χρειάζονται οι πολίτες για να έχουν ασφαλή πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους για να υποστηρίξουμε ακριβώς τους καρκινοπαθείς και τέλος θεραπεία του καρκίνου δεν έχει να κάνει με την απλή επιβίωση. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επανένταξη του κόσμου στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Να είναι όσο γίνεται πιο εύκολη αυτή για τις γυναίκες και ε, φέρουν ευθύνη οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και άλλοι φορείς. Και ε, το Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων θα θυμάστε ότι ε, το συζήτησε το 2018 και τώρα ε, ε, δεν ακούμε τίποτα από τον πρόεδρο ε, την Προεδρία. Θα πρέπει να δείξουμε πολιτική βούληση και να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να κάνουν πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελειώνει η συζήτηση αυτή εδώ. Έχουμε λάβει ένα ψήφισμα για να ψηφιστεί αύριο. Ευχαριστώ. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι κοινή συζήτηση. Ε, και πριν σας αναγνώσω τα θέματα, να γίνει αλλαγή σκητάλης εδώ ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Κοινή συζήτηση για τα δικαιώματα των ε, ΛΟΑΔ με προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα των μεσοφιλικών ατόμων από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Επίσης έχουμε προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑ 2019-2023 ε, από διάφορες πολιτικές ομάδες. Αρχίζει η συζήτηση με από τους συντάκτες ε, των κοινών αυτών ερωτήσεων. Ο κύριος Μωράες, για πέντε λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διακρίσεις κατά τον ΛΟΑΔΜΑ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε εντάξει το ζήτημα αυτό στη σημερινή ημερήσια διάταξη και ότι διεξάγουμε τη σημερινή συζήτηση. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό και θα ήθελα όλου ιδιαίτερω να ευχαριστήσω και την διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ καθότι συνέβαλε και αυτή η ομάδα στο να τεθεί το σημερινό ζήτημα στην μερίσια διάταξη. Θα ήθελα να τονίσω ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά τον ΛΟΑΔΜΑ. Θα ήθελα να πω ότι ε, για πρώτη φορά αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη πτυχή του όλου ζητήματος, καθότι ε, ανάλογη συζήτηση έχει γίνει και στην ΟΕΕ δηλαδή της Ευρώπης, αλλά πρώτη φορά διεξάγεται τέτοια συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εστιαζόμαστε συγκεκριμένα στα μεσοφιλικά άτομα. Συζητάμε λοιπόν το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να επικεντρωθεί η παρέμβασή μου αυτή στο ψήφισμα και το, την προφορική ερώτηση της α, Επιτροπής η οποία ασχολείται με ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν συζητείται πάρα πολύ συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά θέλουμε να αποτιμήσουμε τις αξίες Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με όλου του πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλε τι κοινότητε. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να εστιαστούμε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα μεσοφιλικά άτομα και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω και θα πρέπει να πούμε ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνουν τα μεσοφιλικά άτομα είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει λοιπόν να τις θέσουμε πραγματικά στις προτεραιότητές μας. Τα μεσοφιλικά άτομα αντιμετωπίζουν παραβιάσεις τη σωματική του ακαιρεότητα. Πολλέ φορέ αντιμετωπίζονται ως άτομα τα οποία είναι ασθενή και τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν μια θεραπεία και γι' αυτό το λόγο πολύ συχνά εφαρμόζονται στα άτομα αυτά επεμβάσει χειρουργικέ, επεμβάσεις αποκατάσταση. Ξέρετε ότι τέτοιε επεμβάσει προβλέπονται σε 21 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια τη ζωή του αντιμετωπίζουν στιγματισμό, αρνητική ρητορική, πολλέ φορέ παρενόχληση, επιθέσει και εκφοβισμό στο χώρο εργασία, περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ακόμα και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γενικά ζουν στι κοινωνίε μα εντελώ παραμελημένοι και παραγωνισμένοι. Και πολύ συχνά δεν υπάρχει απαραίτητη νομική τους αναγνώριση. Σήμερα λοιπόν κύριε Επίτροπε καλούμε την Επίτροπη και το, και Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν την παθολογικοποίηση των τόπων αυτών, να, προχωρήσουν στην αποπαθολογικοποίησή τους να καταφέρουν να γλιτώσουν τα άτομα αυτά από τι αναγκαστικέ χειρουργικέ επεμβάσει. Πρόοδο έχει σημειωθεί σε κάποια κρατημέλη, αλλά όχι σε όλα. Θα πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών, να μην είναι θύματα διακριτική μεταχείρισης. Θα πρέπει επίση να έχουν την ε, απαραίτητη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, να μπορεί να γίνεται μια ευέλικτη καταχώρηση του φίλου τους χωρίς να αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα που θέτουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ακόλουθο, τα ακόλουθα μάλλον ερωτήματα. Ξέρω ότι ασχολείται με το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλέ φορέ, μα το έχει πει και στην αρμόδια Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ακόμα μια οριζόντια οδηγία κατά τη διακριτική μεταχείριση που να καλύπτει και τα μεσοφιλικά άτομα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το ακόλουθο. Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο αυτή την οδηγία κατά των διακρίσεων. Έπειτα, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα μεσοφιλικά άτομα, τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά φίλου τους δεν θα αποτελούν σε καμία περίπτωση λόγο διακρατικής μεταχείρισης. Μόνο η Μάλτα και η Πορτογαλία είναι οι χώρες αυτές οι οποίες λένε ότι δεν χρειάζεται οι άνθρωποι αυτοί να υπόκεινται συγκεκριμένε χειρουργικέ επεμβάσει. Και είναι μόνο οι χώρε αυτέ τελικά οι οποίε καταδικάζουν τη διακριτική μεταχείριση μόνο, τον μόνο λόγω των σωματικών χαρακτηριστικών φύλου των ανθρώπων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα λοιπόν να θέσουμε επιτάπητο στο ζήτημα αυτό και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε κοινέ καθολικέ αξίε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίε τις οποίε πραγματικά να προασπιζόμαστε, τότε πραγματικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με τι πιο ευάλωτε ομάδε τη κοινωνία μα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τι περιπτώσει εκκριτική μεταχείρισης και θα πρέπει πραγματικά να ορθώσουμε τον άστημά μα κατά των διακρίσεων αυτών. Γι' αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ περήφανο που μπορούμε και έχουμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την προφορική ερώτηση και το σχετικό ψήφισμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συντάκτες. Στο αρτικό λεξολοάδμα, το μη είναι τα μεσοφιλικά άτομα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την ιδεολογία Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από τις διακρίσεις και τη βία από ε, μικρή ηλικία. Χαίρομαι και είμαι περήφανη που είμαι συντάκτρια της, του πρώτου ψηφίσματος για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ υπάρχουν παιδιά που υπόκεινται σε επεμβάσεις χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και αυτό ζημιώνει την αναπαραγωγική του υγεία. Φανταστείτε αυτό να ήταν το δικό σας παιδί. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού τα ανθρώπινα δικαιώματα υφίστανται επίθεση. Υπάρχει αύξηση της ε, σεξιστική και ξενοφοβική ρητορική και τα ΛΟΑΔΜ άτομα είναι εύκολος ε, στόχος αυτών των διακρίσεων. Δεν θα, ε, δεν έπρεπε να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στη σημερινή κοινωνία και συμφωνώ με τον Κλοντ Μωράες ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων θα πρέπει να προωθηθεί. Είναι απαράδεκτο που παρεμποδίζεται εδώ και χρόνια στο Συμβούλιο. Πολύ συχνά τα άτομα ΛΟΑΔΜ είναι θύματα ε, σχολικού εκφοβισμού, ε, στιγματισμού και διαφόρων άλλων αρνητικών φαινομένων. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ε, ως ευρωπαϊκή κοινωνία και να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς να τους παρέχουμε μια ποιοτική ζωή με αξιοπρέπεια. Η νομοθεσία που ε, προέχει, παρέχει μάλλον ε, την πρόσβαση ε, στην νομική υποστήριξη είναι ένα απαραίτητο βήμα, αλλά δεν πρέπει να είναι το μοναδικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε τον μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα που λύγει τώρα. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφή στρατηγική, ένα σχέδιο δράσης να μεριμνήσει για την ε, προστασία των ε, ατόμων ΛΟΑΔΜ και στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Να αναγνωρίσουμε ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Madam. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπιόρκη για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Τα ΛΟΑΔΜ άτομα υφίστανται διακρίσεις ε, εγκλήματα μίσους, απειλές, οι οικογένειές τους βιώνουν ε, τα ίδια, τα διεμφυλικά άτομα ε, και τα μεσοφυλικά άτομα υφίστανται κακοποίηση, επεμβάσεις αποκατάστασης φύλου πράγματα τα οποία εξακολουθούν να γίνονται τώρα στο 2019. Υπάρχουν βελτιώσεις σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες όμως ε, δρομούμε Και τελικά τα άτομα μου θεωρούν ότι είναι... Ε, κάτι το εξωπραγματικό και ότι δεν είναι φυσιολογική. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε την αλληλεγγύη μας ε, με τα, το κίνημα των ε, queer. Πρέπει να δείξουμε τον ανθρωπισμό μας. Απαιτούμε περισσότερη πολιτική δράση. Δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε ε, σε μερικές μικρές υποχωρήσεις ε, που θέλουμε να καταγραφούν ρητός εξαιτίας του Όρμπαν και άλλων. Χρειαζόμαστε μια πραγματική στρατηγική ε, υπέρ των ΛΟΑΔΜ, κατά, κατά των διακρίσεων, να σταματήσουμε ε, τα εγκλήματα μίσους, πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά ΛΟΑΔΜ ανά την Ευρώπη. Εμείς ε, δεν θα χαθούμε, θα επανέλθω ή σκοπεύω να επανέλθω ως Ευρωβουλευτής μετά τις εκλογές του Μαΐου και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί και το σώμα μας και η ζωή μας, τα όνειρά μας δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα, είναι και μια ευκαιρία να σπάσουμε αυτές τις ε, παραδοσιακές ε, στερεοτυπικές εικόνες για το τι είναι τα άτομα ΛΟΑΔΜ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιώτη για δύο λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τα δύο φτερωτήματα με τα οποία ουσιαστικά θα κλείσει και η εργασία αυτή τη κοινοβουλευτική εντολή, είναι δύο ερωτήματα στα οποία συνέβαλαν πάρα πολλοί συνάδελφοι στα πλαίσια τη διακομματική ομάδα ΛΟΑΔΜΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήθελα πραγματικά να το πω αυτό και το λέω με ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Μέσω λοιπόν του σχετικού ψηφίσματο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΑ θα αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2019 ω το 2024. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια στρατηγική σφαιρική παρακολούθηση σε όλων των δράσεων προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προωθούν περισσότερο τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, λεσβιών, αμφιλοφίλων ομοφύλων, διεμφυλικών και μεσοφιλικών. Θα πρέπει για όλα αυτά τα άτομα να ισχύουν ισότιμα δικαιώματα με του υπόλοιπου Ευρωπαίου πολίτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει δυστυχώ ακόμα την δυνατότητα να αντιμετωπίσει σφαιρικά και οριζόντια την διακριτική μεταχείριση λόγω ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή χαρακτηριστικών του φύλου. Δυστυχώς φαινόμενα τέτοια έχουμε σε πάρα πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν χώρες που απαιτούν πραγματικά τη στήρωση προκειμένου να αναγνωρίσουν νομικά το φύλο ενός ατόμου ή απαιτούν ακόμα και διάγνωση όσον αφορά την ψυχική υγεία ως προϋπόθεση για να αναγνωρίσουν το φύλο ενός ατόμου. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μεσοφιλικά παιδιά τα οποία υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να του ε, καθοριστεί τελικά το ένα ή το άλλο φύλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία σίγουρα δεν τα προστατεύουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Στα πλαίσια του προγραμματισμού λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να καταφέρουμε να προστατεύσουμε όλου του πολίτε από τη διακριτική μεταχείριση μέσω τη οριζόντια αυτή οδηγία που όπω ακούσαμε παρεμποδίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι ε, η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ίδια τα άτομα, ΛΟΑΔΜΑ αλλά και τι οικογένειέ του.